Καλημέρα σε όλους και καλωσορίσατε στη σημερινή συνέντευξη τύπου. Θα αρχίσουμε απευθείας και θα ολοκληρωθεί η συνέντευξη ακριβώς στις 11.30, 10 ε, λεπτά με 15 για μας ε, και 15 με 20 για τους δημοσιογράφους. Η Γκάμπι Τσίμερ, παρακαλώ, θα λάβει πρώτο λόγο. Καλημέρα. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ε, καλωσορίσω. Ε, ήδη πριν από ένα χρόνο η πολιτική μας ομάδα GUNGL είχε καλέσει τον κύριο Τσίπρα, πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, για να έρθει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εκείνη την εποχή ο στόχος ήταν να συζητήσουμε τις ε, συμφωνίες που είχαν συναυθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Σήμερα η επικαιρότητα είναι η άνοδος ε, των φασιστικών τάσεων στην ε, Ευρώπη. Έχουμε ήδη ξεκινήσει στους κόλπους της ομάδας μας μια σχετική συζήτηση. Έχουμε επίσης συζητήσει με τον Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με το βαθμό στον οποίο η σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα μπορεί να επηρεάσει, επηρεάσει συγγνώμη, την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να αγωνίζονται για την απλή τους επιβίωση, είναι απαράδεκτο να συζητάμε για αποπληρωμή χρέους. Υπάρχουν ευθύνες, υπάρχουν ευθύνες που πρέπει να επομιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, χρειαζόμαστε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τους ανθρώπους. Ε, η κατάσταση είναι αβάσταχτη. Αλλιώς μόνο έτσι μπορούμε να μιλήσουμε για αποπληρωμή χρέους ή για την νομιμότητα των χρεών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει... να το αντιληφθεί αυτό. Και ο Επίτροπος και ο Πρόεδρος Μπαρόσο το Σεπτέμβριο με τις ομιλίες τους προέβησαν στην ίδια εκτίμηση ότι είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι μόνο να πιέσουμε το επιμέρους κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του, αλλά να επιδείξει και να θέσουμε στο επίκεντρο της προσοχής την αλληλεγγύη. Αυτό απαιτούν και οι συνθήκες, το θεωρούν αυτονόητο και αυτό που ζητούμε, σε αυτό άλλωστε συζητούμε και με τον Αλέξη Τσίπρα, είναι με ποια μορφή μπορούν οι συνθήκες, το πλέγμα αυτό το νομοθετικό, το κανονιστικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δείξουν την αλληλεγγύη σε μια κατάσταση τόσο δύσκολη στην οποία βρίσκονται οι λαοί. Αυτό είναι το θέμα της συζήτησή μας και αυτό είναι το σημείο εκκίνησης και για τους προσεχείς μήνες. Έτσι λοιπόν χαίρομαι πολύ που μπορώ να καλωσορίσω σήμερα εδώ τον Αλέξη Τσίπρα και του δίνω αμέσως το λόγο. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Ε, βρίσκομαι εδώ μετά από πρόσκληση της ε, Ευρωομάδας της Αριστεράς, QNGL, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να συνομιλήσω ε, με τους Ευρωβουλευτές και τις Ευρωβουλευτίνες της Ομάδας Αριστεράς, αλλά και με την ευκαιρία να συναντηθώ με ε, ηγετικά στελέχη της, του Ευρωκοινοβουλίου και της της Κομισιόν προκειμένου να θέσω για άλλη μια φορά ε, το κρίσιμο ε, ζήτημα της ε, αδυναμίας του προγράμματος που εφαρμόζεται στην Ελλάδα από την Τρόικα εδώ και τρία σχεδόν χρόνια να ανταποκριθεί στοιχειοδός στους οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους. Και θέλω να είμαι πολύ σύντομος στην εισαγωγή μου για να δώσω τη δυνατότητα να, να, να ρωτήσετε και να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Θα σας πω λοιπόν ότι Ήρθε η στιγμή για τους Ευρωπαίους πολιτικούς να αντιμετωπίσουν την αλήθεια σε σχέση με, το πρόγραμμα ε, του μνημονίου, το οικονομικό πρόγραμμα στην Ελλάδα αλλά και συνολικά στους, ε, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας. Ήρθε η στιγμή να αντιμετωπίσουν ε, κατάματα τους Ευρωπαίους φορολογούμενους, Ευρωπαίους πολίτες και να δώσουν απαντήσεις. Οι γερμανικές εκλογές τελείωσαν. Δεν υπάρχουν λοιπόν ε, σκοπιμότητες πια. Πρέπει να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Και η γλώσσα της αλήθειας είναι ότι αυτό που εδώ και τρία χρόνια εφαρμόζεται στην Ελλάδα είναι ένα αδιέξοδο πρόγραμμα που έχει οδηγήσει την ελληνική κοινωνία στα πρόθυρα ανθρωπιστικής κρίσης. Ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έχει πιάσει κανέναν από τους στόχους του και πολύ δε περισσότερο ένα πρόγραμμα το οποίο αν συνεχίζει να εφαρμόζεται εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για την ίδια τη συνοχή της, Ευρωζών, της, Ευρω... της Ευρωζώνης και της Ευρώπης. Η κίνδυνη είναι διτή Πρώτον, ε, η ανθρωπιστική κρίση την οποία σας περιέγραψα Ήδη έχουμε ε, αποτελέσματα τα οποία είναι συγκλονιστικά. Η ανεργία στην Ελλάδα, η επίσημη καταγεγραμμένη ανεργία έχει ε, προσεγγίσει το 30%. τους νέους ανθρώπους υπερβαίνει το 60%. Το 1 τρίτο του πληθυσμού ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας. Υπάρχει διάχυτη στην κοινωνία αίσθηση αδικίας Υπάρχει διάχυτη στην κοινωνία αίσθηση οργής. Αυτό αυτομάτως καταγράφεται και σε υψηλά ποσοστά σκεπτικισμού σε σχέση με την Ευρώπη και το μέλλον της. Και την ίδια στιγμή έχουμε ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο, το κίνδυνο της επόασης, της ανάπτυξης του φασισμού στην Ελλάδα. Είχαμε μια θετική εξέλιξη σε ό,τι αφορά την σύλληψη και την, ε, τη, ε, τη, σύλληψη και την εξάρθρωση της εγκληματικής δραστηριότητας της Χρυσής Αυγής. Εν τούτης όμως το φαινόμενο της ανάπτυξης του φασισμού συνεχίζει να μας απειλεί και σε μεγάλο βαθμό έχει να κάνει, οι αιτίες δηλαδή που τον προκαλούν είναι ε, οι νεοφιλελεύθερες, σκληρές, βάρβαρες οικονομικές πολιτικές λιτότητας. Και αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αυτό είναι μια απειλή για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, είναι μια απειλή για την Ευρώπη. Ως εκ τούτου λοιπόν ε, είμαστε εδώ για να θέσουμε για άλλη μια φορά στην ε, ευρωπαϊκή ηγεσία το αίτημα να μιλήσουν με τη γλώσσα της αλήθειας απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες, στους Ευρωπαίους φορολογούμενους για το ελληνικό πρόβλημα που δεν είναι ελληνικό, είναι ευρωπαϊκό δηλαδή να μιλήσουν για το ευρωπαϊκό πρόβλημα. Η απάντηση λοιπόν στο ευρωπαϊκό πρόβλημα δεν είναι η λιτότητα. Όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα αυτό το χρέος μας ήταν στο 110% του ΑΕΠ, σήμερα είναι στο 170% του ΑΕΠ. Η απάντηση δεν είναι η περιοριστική πολιτική. Το μνημόνιο δεν μπορεί να συνεχίζει να εφαρμόζεται διότι παράγει αδιέξοδα. Και αυτό δεν αφορά μόνο μια επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ αφορά μια ε, συζήτηση που πρέπει να γίνει ε, στο υψηλότερο δυνατό ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι ακόμα και αν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ελληνικός λαός που έλεγε ως εδώ, δεν πάει παραπάνω, δεν αντέχουμε άλλα μέτρα λιτότητας, ε, η ίδια η ευρωπαϊκή ηγεσία θα έπρεπε να αναστοχαστεί και να δώσει απαντήσεις για το πώς θα μπορέσει να συνεχίσει την υλοποίηση ενός οικονομικού προγράμματος αδιέξοδου πάνω σε κοινωνικά ερήπια. Μας λένε ότι ε, θα πρέπει μέχρι το 2020 να έχουμε πλεονάσματα της τάξης του 4,5% του ΑΕΠ, πρωτογενή πλεονάσματα, προκειμένου να μπορούμε να αποπληρώσουμε, να μπορέσουμε να αποπληρώσουμε ε, τόκους και χρεολύσια που φτάνουν περίπου στα 83 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2020. Αυτό είναι πρακτικά ανέφικτο για μια χώρα που βρίσκεται για έκτη συνεχόμενη χρονιά στην ύφεση, έχει χάσει το 25% το καθάριστο εγχώριου προϊόντος της και δεν υπάρχει καμία αισιόδοξη προοπτική ότι το επόμενο διάστημα, παρά τις προβλέψεις αρχικές, δεν υπάρχει καμία αισιόδοξη προοπτική ότι θα μπορέσουμε να ανακάμψουμε. Άρα λοιπόν ε, εδώ δεν είναι ζήτημα, επιτρέψτε μου, ιδεολογίας ή ιδεολογικής προσέγγισης. Είναι ένα πραγματικό πρόβλημα, πρέπει να δοθούν απαντήσεις, πρακτικές απαντήσεις και πρέπει η ευρωπαϊκή ηγεσία να τεθεί μπροστά στις μεγάλες ευθύνες που την, ε, ε, πολύ μεγάλες ευθύνε που έχει δεδομένου ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας γενικευμένης κοινωνικής, πολιτικής κρίσης και κοινωνικής κρίσης. Η εξάπλωση του φασισμού είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, είναι ένα κίνδυνο για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Η διάλυση της κοινωνικής συνοχής στην Ελλάδα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, είναι ένα κίνδυνο για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Άρα λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι ήρθε η στιγμή να πάψουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η λύση που προτείνουμε, και κλείνω με αυτό, για να δώσω τη δυνατότητα σε όλους να απευθύνετε τις ερωτήσεις σας. Η ευρωπαϊκή λύση που προτείνουμε αφορά ε, μια ε, διάσκεψη ευρωπαϊκή για το χρέος προκειμένου να ε, βρεθεί μέσα από τη διαγραφή μεγάλου μέρους του, μέσα από μορατόριουμ στην αποπληρωμή των τόκων και ρήτρα ανάπτυξης που θα αφορά βεβαίως όχι μόνο την Ελλάδα αλλά όλες τις χώρες της περιφέρειας που αντιμετωπίζουν ε, παρόμοιο πρόβλημα, να βρεθεί μια βιώσιμη λύση που θα δίνει προοπτική, που θα δώσει τη δυνατότητα στις χώρες αυτές, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, να μπορέσουν να ξαναβγούν στις αγορές και να πάψουν να χρεώνουν τους Ευρωπαίους φορολογούμενους. Η λύση που προτείνουμε εμπεριέχει το, την ε, ε, αναπτυξιακή χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων των ε, χωρών της περιφέρειας προκειμένου να καταπολεμήσουμε τον, ε, την ε, διόγκωση της ανεργίας, την αύξηση της ανεργίας, να υπάρξει ανάπτυξη η οποία θα μπορέσει να ξαναφέρει τις χώρες αυτές σε τροχιά κοινωνική συνοχής. Η λύση που προτείνουμε είναι το βάθεμα της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Και εν ώψη των ευρωπαϊκών εκλογών οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι οι επιλογές που έγιναν πρώτα με την Ελλάδα, ακολούθως και στις υπόλοιπες χώρες της ε, ε, Ευρωπαϊκής Περιφέρειας, του Ευρωπαϊκού Νότου, ήταν επιλογές που συρρήκνωσαν τη δημοκρατία, ε, μη αιρετοί, μη εκλεγμένοι οργανισμοί παίρνουν αποφάσεις για τους λαούς ερήμην των λαών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να συνεχίσει να έχει έναν ρόλο ε, ούτε καν συμβουλευτικό, ένα ρόλο θεατή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει κυρίαρχο ρόλο, οι λαοί πρέπει να έχουν κυρίαρχο ρόλο για το μέλλον τους, για το μέλλον της Ευρώπης. Η παρουσία μας λοιπόν εδώ είναι μια κραυγή αγωνίας για τις εξελίξεις στην Ελλάδα, μια κραυγή αγωνίας για το μέλλον της Ευρώπης που πραγματικά ε, ε, είναι δυσίωνο αν συνεχιστούν αυτές οι επιλογές, αλλά και μια τοποθέτηση ρεαλισμού και ευθύνης για το ποιε μπορεί να είναι οι ενδεδειγμένες λύσεις μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, ώστε να υπάρξει διόρθωση των αστοχιών, ώστε να υπάρξει ε, ξανά τροχιά ανάπτυξης και συνοχής στην ε, ευρωπαϊκή περιφέρεια και συνολικά στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Με αυτές τις σκέψεις είμαι στη διάθεσή σας για ε, τις απαντήσεις στα ερωτήματά σας. Παρακαλώ. Νίκος Χρυσολαράς από την Καθημερινή. Ήθελα να ρωτήσω την κυρία Τζίμερ αν ε, εν ώψη των ευρωπαϊκών εκλογών ε, το, το κόμμα της αριστεράς θα έχει ε, ενιαίο υποψήφιο για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν συζητείτε το όνομα του κυρίου Τσίπρα για, για, υπο, για την υποψηφιότητα αυτή και θα ήθελα να ρωτήσω και τον κύριο Τσίπρα αν ενδιαφέρεται να είναι υποψήφιος με το κόμμα της αριστεράς για την Προεδρία της Κομισιόν. Για την ερώτησή σας θα σας απαντήσω ότι εδώ βρίσκομαι ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας GUE NGL. Δεν είναι πολιτική ομάδα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Ως αυτό από τη θέση την οποία εκπροσωπώ εδώ δεν μπορώ να δώσω απάντηση στο ερώτημά σας διότι συμμετέχουν στην πολιτική ομάδα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κόμματα τα οποία δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Αριστερά. Ωστόσο είμαι και μέλος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και ως ιδιώτης μπορώ να σας απαντήσω ότι το Δεκέμβριο η Ευρωπαϊκή Αριστερά είχε ένα συνέδριο στη Μαδρίτη στη, διάρκεια του οποίου θα ληφθεί η απόφαση φυσικά με ψηφοφορία για το πώς θα ταχθεί στο θέμα των ευρωεκλογών και ως ιδιώτης θα ήθελα επίσης να σας πω ότι θα μου φαινόταν πάρα πολύ ωραίο, καταπληκτικό το να έχουμε στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα ένα έναν πολιτικό Ευρωπαίο εφόσον ενδιαφέρεται να ε, τεθεί επικεφαλής της προτάσεως της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Αυτό το λέω ως ιδιώτης γιατί δεν μπορώ να εκπροσωπήσω κόμματα τα οποία δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Αριστερά και βρίσκονται στην ίδια πολιτική ομάδα στο Κοινοβούλιο. Στο ίδιο μήκο να σας πω με ευθύτητα ότι δεν ε, αποτελεί μέρος της ε, ατζέντα των συζητήσεών μας το θέμα που θέσατε διότι όπως πολύ καλά γνωρίζετε οι αποφάσεις θα παρθούν πρωτίστως σε επίπεδο κομμάτων και βεβαίως ε, δευτερευόντως ε, θα υποστηριχθούν αυτές οι αποφάσεις από τις ε, ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άρα δεν αποτέλεσε αντικείμενο παρά τις αντίθετες φήμες που διάβαζα και εγώ στον ελληνικό τύπο δεν αποτέλεσε αντικείμενο της επίσκεψής μου το θέμα αυτό. Σε ό,τι αφορά την ουσία του ερωτήματο, εγώ θέλω να σας πω. Ε, εμάς μας ενδιαφέρει η δυνατότητα που υπάρχει η Ευρωπαϊκή Αριστερά να έχει το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε αυτές τις ευρωπαϊκές εκλογές. Αυτό μας ενδιαφέρει και ως Έλληνες αριστερούς και ως Ευρωπαίους αριστερούς. Αυτό απαιτεί ενότητα, στρατηγική, σχέδιο, πολιτικό πρόταγμα. Τα πρόσωπα δεν έχουν αμεληταίο ρόλο, αλλά πρωτίστως σημασία έχει το πρόγραμμα, η στρατηγική και η ευρύτερη δυνατή ενότητα. Μας ενδιαφέρει αυτό και για ένα λόγο παραπάνω εμάς τους Έλληνες αριστερούς. Διότι πιστεύουμε ότι η άνοδος των ε, προοδευτικών, των αριστερών δυνάμεων στην ε, Ευρώπη και στις επικείμενες ευρωεκλογές μπορεί να αποτελέσει το κατάλληλο έδαφος για να μπορέσουμε να πετύχουμε και εμείς μια σημαντική εκλογική νίκη στην Ελλάδα και να αλλάξει ριζικά το κλίμα και οι συσχετισμοί στην Ευρώπη ώστε η Ευρώπη να μπορέσει ε, να αντιμετωπίσει την ουσία των προβλημάτων χωρίς ε, δαιμονοποιήσεις και να μπορέσει να δεχτεί ότι μια ε, αριστερή κυβέρνηση που δημοκρατικά θα εκλεγεί στην Ελλάδα θα συμβάλλει στην ε, ε, αλλαγή στρατηγική συνολικά προς όφελος όλων των ευρωπαϊκών λαών, διότι εμείς δεν αντιμετωπίζουμε την, ε, την διαπραγμάτευση ή τη σύγκρουση που θα υπάρξει, τη σύγκρουση απόψεων για το μέλλον της Ευρώπης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μετά την εκλογή μιας αριστερής κυβέρνησης στην Ελλάδα, ως μια αντιπαράθεση ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς λαούς, αλλά ως μια πολιτική αντιπαράθεση, ανάμεσα στρατηγικέ. στρατηγικές. Και θέλω να επισημάνω ότι η δική μας στρατηγική, η στρατηγική δηλαδή της κοινωνικής σωτηρίας στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας, είναι μια φιλοευρωπαϊκή στρατηγική. Αντιθέτως, η στρατηγική που σήμερα ακολουθείται από τις συντηρητικές ηγεσίες στην Ευρώπη είναι μια αντιευρωπαϊκή στρατηγική. Uh, Μία επερώτηση. Ο κύριος Τσίπρας δεν ξεκαθάρισε στην παρέμβασή του αν προτίθεται να καταθέσει υποψηφιότητα ή όχι. Στο μέτρο βεβαίως που η πλειοψηφία της ομάδας θα στο ζητήσει να είστε υποψήφιος. Ε, εν τη αυτή περιπτώσει θα το δεχόσασταν. Επίσης, μπορείτε να διευκρινίσετε περαιτέρω την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Αριστεράς για την αντιμετώπιση της κρίσης. <laughs> Στην Ελλάδα έχουμε μια ε, παροιμία που ε, λέει κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολλιός που είναι ένα πολύ ε, εύγευστο ψάρι τον Αύγουστο. <laughs> <laughs> Λοιπόν, δεν είναι η ώρα να σας απαντήσω σε αυτά τα ερωτήματα τα οποία, για τα οποία θα ασχοληθούν ε, ε, συλλογικά όργανα. Διότι όπως πολύ καλά γνωρίζετε εμείς στην αριστερά λειτουργούμε μέσα από συλλογικέ διαδικασίες και παίρνουμε συλλογικές αποφάσεις. Ε, στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας σε σχέση με τη στρατηγική της αριστεράς. Νομίζω ότι η αριστερά στην Ευρώπη είναι η πολιτική δύναμη που με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο από την πρώτη στιγμή διατύπωσε την άποψη ότι τα προγράμματα της λιτότητας όχι μόνο είναι αναποτελεσματικά αλλά είναι καταστροφικά. Όχι μόνο οδηγούν σε ε, συνθήκες ε, βαρβαρότητας ε, και διαρριγνύουν την κοινωνική συνοχή αλλά δεν θα έχουν και κανένα αποτέλεσμα σε σχέση με το οικονομικό πρόβλημα που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Και νομίζω ότι η αριστερά δικαιώθηκε για αυτή τη στάση. Και ήταν η μόνη πολιτική δύναμη και η μόνη ομάδα που το έθεσε αυτό με απόλυτη σαφήνεια και που έθεσε και αντιπροτάσεις. Δεν κατήγγειλε μόνο την ακολουθούμενη πολιτική, αλλά έθεσε και προτάσεις ώστε μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο να υπάρξει μια εναλλακτική πολιτική η οποία θα είναι αποτελεσματική και βιώσιμη. Θέλω να πω ότι ε, οι δύο κορυφαίες ε, ε πολιτικές οικογένειες ε, επέλεξαν, ενώ η οικογένεια της λαϊκής δεξιάς και η σοσιαλδημοκρατική, με τον ένα τον άλλο τρόπο είτε επέλεξαν είτε ανέχτηκαν πολιτικές που και οι ίδιοι γνωρίζανε ότι στο τέλος θα δικήσουν αδιέξοδο. Και σήμερα βρίσκονται και οι ίδιες μπροστά σε αυτό το στρατηγικό αδιέξοδο. Ως εκ τούτου, με τη στρατηγική της υπέρβασης της λιτότητας, με τη στρατηγική της ε, ε, ενίσχυσης της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής, θα προσέλθουμε, ε, θέλω να πιστεύω, με την ευρύτερη δυνατή ενότητα δυνάμεων σε αυτές τις ευρωεκλογέ, ελπίζοντας ότι πράγματι θα έχουμε ένα άλμα στην ε, εκπροσώπησή μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είδαμε πάρα πολλές αλλαγές ως προς την τακτική ή τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Πιστεύετε ότι ενδέχεται να τροποποιηθεί η πολιτική λιτότητα ε, εάν δεν είναι εντελώς διαφορετική σύνθεση του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεύτερον έχετε ελπίδες για την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύουμε ότι μετά από τρία χρόνια της Ελλάδας στο μνημόνιο και μετά από αρκετά χρόνια όπου κυριαρχούν τα δόγματα, τα νεοφιλελεύθερα της λιτότητας ε, σε όλη την Ευρώπη, τα ίδια τα αποτελέσματα και η ίδια η ζωή έχει δείξει ε, ότι ε, δεν οδηγούμαστε πουθενά. Άρα λοιπόν οι ελπίδες μου δεν έχουν να κάνουν με το ότι οι ίδιοι άνθρωποι θα αλλάξουν ιδέες ή θα αλλάξουν απόψεις, αλλά με το ότι η ίδια η ζωή μας βάζει μπροστά σε αποφάσεις. Ο κόμπος έχει φτάσει στο κτένι. Είναι αναγκασμένη η ευρωπαϊκή ηγεσία να πάρει αποφάσεις, ιδαλλιώς θα βρεθούμε πολύ γρήγορα μπροστά σε αδιέξοδα που θα αφοράν το ίδιο το μέλλον και την ίδια τη συνοχή της Ευρώπης. Εκτιμώ λοιπόν ότι πολύ σύντομα θα ανοίξει αυτή η συζήτηση με αφορμή το ελληνικό πρόβλημα, την, ε, την ε, ε, αστοχία του προγράμματος στην Ελλάδα, την πλήρη αστοχία του προγράμματος στην Ελλάδα, αλλά θα ανοίξει και διότι ε, και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ε, και στις υπόλοιπες χώρες της περιφέρειας και του Νότου έχουμε και κοινωνική κρίση και πολιτική κρίση και οικονομικά διέξοδα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα αναγκαστεί η ευρωπαϊκή ηγεσία σε αλλαγή προσανατολισμού και σε διορθώσεις. Εάν το ε, αποτέλεσμα των εκλογικών αναμετρήσεων και στις ε, ε, χώρες ξεχωριστά αλλά ιδιαίτερα στις ευρωπαϊκές εκλογές δώσει και ένα ισχυρό μήνυμα αλλαγής, νομίζω ότι τότε θα μπορούμε να μιλάμε και να ελπίζουμε για αλλαγή πορείας. Σε σχέση με την ελληνική προεδρία πρέπει να σας πω ότι δεν περιμένουμε πολλά. Δεν περιμένουμε πολλά δεδομένου ότι ε, η ελληνική κυβέρνηση έρχεται απροετοίμαστη για ένα σημαντικό γεγονός α, αρκούμενη στη δικαιολογία ότι μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας οι προεδρίες των χωρών δεν παίζουν και τόσο πολύ σημαντικό ρόλο. Εμείς παρόλα αυτά είμαστε προετοιμασμένοι. Διότι όπως γνωρίζετε η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα είναι ρευστή και ανα πάσα στιγμή, εμείς το διεκδικούμε άλλωστε, μπορεί να προκηρυχθούν προώρες εκλογές. Και έχουμε εξετάσει και έχουμε δουλέψει στο ενδεχόμενο η ελληνική προεδρία να γίνει με μια κυβέρνηση της αριστεράς στην Ελλάδα. Και έχουμε προετοιμαστεί για αυτό το ενδεχόμενο, ώστε εάν συμβεί, να είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία που δεν θα χάσουμε, θα δράξουμε την ευκαιρία ώστε να θέσουμε τα πραγματικά διλήμματα και τα πραγματικά προβλήματα που αφορούν τη βιωσιμότητα, την προοπτική, το μέλλον της Ευρώπης και των λαών της. Θα ήθελα σύντομα να προσθέσω και εγώ από τη δική μου έποψη Αναφερθήκατε στα τελευταία τέσσερα χρόνια και είπατε αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να επηρεάσει, να επιδράσει σε αυτήν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή αν θα πρέπει να περιμένουμε τη σύνθεση της επόμενη Επιτροπής. Θα σα απαντήσω απλά. Έχουμε επιδράσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για κοιτάξτε τι λέει τώρα ο Μπαρόσο και κάποιοι άλλοι τι τελευταίε ημέρε, το, από το Σεπτέμβριο ήδη. Καταρχά διαπιστώνουν ότι η πολιτική που αξιοποιήθηκε μέχρι τώρα για την αντιμετώπιση της κρίσης έχει αποτύχει, δεν είναι επαρκής. Και δεύτερον, προσανατολίζονται πολύ περισσότερο στο να αναλάβουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση την ευθύνη μας και να επιδείξουμε αλληλεγγύη προς τα κράτη-μέλη. Αυτή η αλλαγή προσανατολισμού λοιπόν προς την απαραίτητη ευρωπαϊκή αλληλέγγυα πολιτική συνοχής. Διαπιστώνουμε τώρα. Στο βαθμό αυτό λοιπόν σας λέγω ναι, είναι δυνατόν, ναι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει να δώσει απαντήσεις, μπορούμε ακόμα να πραγματοποιήσουμε βήματα για να θέσουμε σε κίνηση κάποια πράγματα, αλλά θα σας απαντήσω ξεκάθαρα ότι ο αντισυμβαλόμενος του ΣΥΠΗΝ δεν είναι η Επιτροπή, είναι το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο είναι αυτό το οποίο χαράει στην πολιτική και εκεί ορίζονται οι βάσεις ή εκεί έχουν υπονομευθεί καλύτερα οι βάσεις για την αλληλέγγυα πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον προϋπολογισμό για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο στα διαφορετικά ταμεία βλέπουμε ότι υπονομεύει την κοινωνική πολιτική. Ε, κάποια πράγματα συμπληρωματικά σε αυτά που υπόθηκαν στο, στον πυρήνα της ερώτησης. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ, αλλά και κάποιες επεξηγηματικές περισσότερο ο, ε, για τους λόγους της επίσκεψη Το εξήγησε ο ο σύντροφος, ο πρόεδρος, ο Αλέξης Τσίπρας, με την έκκληση τουλάχιστον στους Έλληνες, αλλά όχι μόνο, και στους άλλους δημοσιογράφους είστε εδώ, ε, με μεγαλύτερη, θα έλεγα, προσοχή και αυστηρότητα, παρακολουθήστε ορισμένες εξελίξεις και τη στάση της Γκουε και τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ σε ευρωπαϊκά θέματα. Παράδειγμα πρώτο, απάντηση. Όταν λέγαμε το έλεγε η Γκουε, το λέγαμε εμείς, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι ο μόνος ερετό θεσμός, πρέπει να ασκήσει τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητές του. Και το κάναμε πολύ συγκεκριμένο. Τι λέει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το μνημόνιο και την Τρόικα που πρώτη φορά εφαρμόστηκε στην Ελλάδα, δεν μας άκουγε κανένας. Ε, το κάτι γραφικό ή και χαρακτηριστικό. Σε τελευταία συνέντευξη, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον οποίο ευχαριστούμε και δημοσίως διότι έχει μια ανοιχτή πρόσκληση για συζήτηση μαζί μας, παραδέχτηκε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ελέγχει τουλάχιστον τα δύο τρίτα της Τρόικα, πρέπει να ελέγξει τα μνημόνια, αν είναι συμβατά με την κοινοτική νομοθεσία. Υπογράμμιση. Θα σας παρακαλούσα να την παρακολουθήσετε αυτή τη διαδικασία. Εμείς αισθανόμαστε δικαιωμένοι και όσοι έλεγαν ότι αυτό το πράγμα είναι έξω από την κοινοτική νομοθεσία, πέρα από όλα τα άλλα που υπόθηκαν. Το δεύτερο Είπαμε ότι δεν είναι μονόδρομοι. Ερχόμαστε εδώ για άλλη μια φορά για να συζητήσουμε με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Κομισιόν, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για να δώσουμε μια απάντηση και έχει σχέση με τις επίκαιρες πολιτικές εξελίξεις, ότι κάναν λάθος όταν στις εκλογές τις προηγούμενες κορυφαίοι θεσμικοί παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούσαν τον ελληνικό λαό να μην ψηφίσει ακραία κόμματα. Θυμόσαστε τις δηλώσεις του κυρίου Γιούγκερ. Θυμόσαστε τις δηλώσεις του κυρίου Ρεν. Θεωρώντας μέσα εκεί ακραία κόμματα τη Χρυσή Αυγή, τις ξέρουμε τις εξελίξεις, αλλά και το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα το σχολιάσω περισσότερο, ξέρετε τις εξελίξεις. Με αυτούς λοιπόν εμείς θέλουμε να τους πούμε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και πρέπει να τις κουβεντιάσουμε. Και δεν έχουν λόγο να αντιμετωπίζουν το ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά με αυτόν τον τρόπο. Αυτά θα ήθελα να προσθέσω ως επιπρόσθετα σχόλια για να μην σας κουράζω περισσότερο και ξαναλέω εξηγεί και το πρόγραμμά μας, εξηγεί και τις προτεραιότητές μας και εδώ είμαστε να απαντήσουμε και σε άλλα ο Πρόεδρος και η Πρόεδρος. Τελευταία ερώτηση. Αθανασίου από το Star και την ε, Real News. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σα ρωτήσω τι θα συζητήσετε καταρχήν με τον Επίτροπο Λάσλο Άντορ και επιπλέον γιατί δεν βλέπετε τον Όλυ Ρεν σήμερα, μια και είστε εδώ. Ναι, ο κύριος Ρεν ε, μου έδωσε ένα ραντεβού χθες το μεσημέρι, αλλά ήταν αδύνατον εγώ να έρθω χθες το μεσημέρι, διότι όπως καταλαβαίνετε δεν μπορώ να λείπω για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από την Ελλάδα σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για τα ελληνικά πολιτικά πράγματα. Ξέρετε, οι εξελίξει είναι καταιγιστικές και ήδη το πρόγραμμά μου στι Βρυξέλλες είναι ε, πολύ μακρύ. Μένω δύο βραδιές και αυτό είναι μεγάλη πολυτέλεια, στο πω έτσι. Ε, θα έχω την ευκαιρία όμως να συναντήσω τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον, ε, να έχω επαφή και με τον πρόεδρο της ομάδας των σοσιαλιστών, αλλά και με τον επίτροπο τον κύριο Λάσλο. νομίζω ότι θα ξέρετε ότι ο ίδιος έχει κάνει πολύ ενδιαφέρουσες δηλώσεις. Μία εξ αυτών αφορούσε την ε, εκτίμησή του ότι το ε, ελληνικό χρέος ε, πρέπει να αναδιαρθρωθεί. Ότι πρέπει να γίνει κούρεμα του ελληνικού χρέους για να μπορέσει να γίνει βιώσιμο. Ως εκ τούτου αντιλαμβάνεστε έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συνάντηση μαζί του. Αντιλαμβάνεστε ότι οι προτάσεις και οι θέσεις μας δεν είναι ερετικές, εκτός πλαισίου. Είναι προτάσεις και θέσεις ρεαλιστικές, βιώσιμες, Χαιρόμαστε να βλέπουμε ότι υπάρχουν και ε, εκπρόσωποι ε, θεσμικών οργάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορεί να έχουμε διαφορετική ιδεολογική αφετηρία που παρόλα αυτά μπορεί να έχουμε σύμπτωση σε επιμέρους ε, θέσεις, κρίσιμες όμως θέσεις για το μέλλον της Ελλάδας και της Ευρώπης. Ως εκ τούτου η συνάντηση και η συζήτηση μαζί του νομίζω θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι ε, είναι και επίτροπος για τα θέματα της εργασίας και αντιλαμβάνεστε ότι μια χώρα με 30% ανεργία, 60% στους νέους και μια χώρα που έχει διαλύσει την, την, εργασιακή της νομοθεσία υπαγόρευση μάλιστα ε, ευρωπαϊκών ε, οργάνων, εξωθεσμικών μεν αλλά οργάνων όπως η Τρόικα, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για μας. Και επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξετάσουμε το κατά πόσο ε, αυτές οι αποφάσεις που ελήφθησαν για τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων και του νομικού πλαισίου των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα συνάδουν με τον ευρωπαϊκό πλαίσιο, το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο. Άρα νομίζω θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ συζήτηση που θα έχουμε μαζί του. Ε, Αναφερθήκατε στι θετικέ εξελίξει με τη σύλληψη μελών τη Χρυσή Αυγή και την εξάρθρωση αυτή τη εγκληματική οργάνωση. Πώ σχολιάζετε όμω το γεγονό ότι ορισμένα από αυτά τα στελέχη βρέθηκαν ελεύθερα. Ευχαριστώ. Κύριε Μύρη, είναι μια είδηση τη τελευταία στιγμή. Ε, θα μου επιτρέψετε πριν ε, προβώ σε οποιοδήποτε σχόλιο να έχω την ε, ε, καλύτερη δυνατή ενημέρωση που δεν την έχω αυτή τη στιγμή, διότι όπως καταλαβαίνετε είναι μια είδηση που την έμαθα λίγο πριν μπω στη, στην αίθουσα για τη συνέντευξη. Ε, Παρ' όλα αυτά, εγώ αυτό που ε, θέλω να επισημάνω, αυτά που θέλω να επισημάνω είναι δύο πράγματα. Πρώτο, για μας δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Χρυσή Αυγή δεν είναι απλά ένα ε, φασιστικό πολιτικό κόμμα, αλλά μια εγκληματική οργάνωση που δρά όχι τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά από το 1987. Και ε, θύματα της δράσης της ε, το γνωρίζετε καλά, ε, ήμασταν πολλές φορές εμείς, οι ιδέες μας, οι σύντροφοί μας, τα μέλη μας, όλα αυτά τα χρόνια. Ε, από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στους θεσμούς, έχουμε εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη και πιστεύουμε ότι θα κινηθεί πέρα και έξω από σκοπιμότητες. Και επιπλέον ανεξάρτητα με την εξέλιξη της ε, δικαστικής ε, ε, έρευνας, εμείς θεωρούμε ότι η προσπάθεια να απομονωθεί και να εξαρθρωθεί, αν θέλετε, το ναζιστικό εξάμβλωμα δεν αφορά μόνο τη δικαιοσύνη και τις κατασταλτικούς μηχανισμούς. Είναι και μία, αν θέλετε, πρωτίστως ιδεολογική, πολιτική και ηθική μάχη την οποία, έχουμε μπροστά μας να δώσουμε και εμείς σε αυτή τη μάχη θα πρωτοστατήσουμε. Δεν έχω περιθώριο να ακούσω άλλες ερωτήσεις. Έχουμε ήδη ξεπεράσει το χρόνο που είχαμε προβλέψει. Μάλιστα, καλά. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους διερμηνείς που θα κάτσουν περισσότερο. Ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ε, εκπροσωπείτε, αν θέλετε, ένα ιστορικό ρεύμα ε, το οποίο έχει πολλές εμπειρίες. Η εμπειρία του από τη δεκαετία του 30 ήταν ότι φυσικά έφταιγε η μεγάλη ύφεση για την ανάπτυξη του φασισμού, έφταιγε όμως και κάτι άλλο. Έφταιγε το γεγονός ότι το ιστορικό αριστερό ρεύμα δεν μπορούσε να ήταν ενωμένο. Έφταιγαν οι θεωρίες της Τρίτης Διεθνούς περί σοσιαλφασισμού και άλλα τέτοια. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν σήμερα αισθάνεστε ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος να διαπράξετε το ίδιο λάθος που έκαναν κάποιοι εκείνη την εποχή μπροστά στο φασιστικό κίνδυνο. Δηλαδή να υποτιμήσετε τη σημασία της ενότητας της αριστεράς για να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα. Θα ήθελα επίσης να ρωτήσω την κυρία Ζήμερ εάν ε, με δεδομένο τις αυτές τις ευρωεκλογές ε, για πρώτη φορά υπάρχει συνθήκη Λισαβόνας που λέει ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής πρέπει κατά κάποιο τρόπο να απηχεί τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών εάν με αυτό δεδομένο θεωρείται ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια σύμπραξη με τις δυνάμεις πέραν του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ώστε μετά από 10 χρόνια να πάψει να έχει η Ευρώπη έναν πρόεδρο επιτροπής που προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ. πολύ σύντομα και βεβαίως υπάρχει η δυνατότητα αλλάζουν οι σχέσεις και οι συσχετισμοί δυνάμεων στην Ευρώπη. Θα το δούμε αυτό τους προσεχείς μήνες, αλλά εμείς ως Ευρωπαϊκό Αριστερό Κόμμα, οπωσδήποτε, μέχρι το Δεκέμβριο θα ορίσουμε τη θέση μας για το πώς θα σταθούμε για να έχουμε έναν υποψήφιο, μία υποψήφιο για την Ευρωπαϊκή Αριστερά και βεβαίως θα προσδιορίσουμε και τη στρατηγική μας για τις ευρωεκλογές και τις προτάσεις μας για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, Ευρωπαϊκή Έννοια, επί τη βάση βέβαια και των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών. Βεβαίω και ενδέχεται, ή θεωρώ μάλλον αρκετά πιθανό ή αυτονόητο να εκλεγούν ε, άλλοι υποψήφοι από αυτού που προτείνουμε εμεί συντηρητικοί παραδείγματα, αλλά εμεί θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Κύριε Σμιθουράκη, με την περίοδο στην οποία αναφέρεστε με την περίοδο της Βαϊμάρης υπάρχουν ομοιότητες αλλά και διαφορές. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να σας πω ότι όλοι πρέπει να ε, γίνουμε σοφότεροι και να πάρουμε μαθήματα από την ιστορία μας και να ε, αξιοποιούμε τη συλλογική μας μνήμη. Ε, είναι σημαντικό να συμφωνήσουμε όμως ότι μία από τις βασικές αιτίες που ανέδειξαν το έκτρωμα του φασισμού στην Ευρώπη και τότε και τώρα είναι οι βάρβαρες οικονομικές πολιτικές. Άρα, ε, αν ε, αυτό αποτελεί την πρώτη προσέγγιση, είναι κάτι που αφορά πρωτίστως την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πρέπει να καταλάβει ότι οφείλει, έχει την ιστορική ευθύνη απέναντι στους λαούς της Ευρώπης να διορθώσει το λάθος που κάνει όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα. Στο δεύτερο που θέσατε εγώ θέλω να σας πω ότι η ελληνική αριστερά ε, έχει ένα άλλο παράδειγμα, πιο πρόσφατο από τη δεκαετία του 30, που ήταν το πώς απάντησε στο φασισμό και στην επέλαση του φασισμού στη χώρα μας τη δεκαετία του 40. Όταν προέταξε το αντιφασιστικό μέτωπο για κάτω από πάρα πολύ σκληρές και αντίξωες συνθήκες. Άρα λοιπόν ε, εμείς ε, έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές με άλλες ε, δυνάμεις ε, στη χώρα μας, ριζικές διαφορές ό,τι αφορά την οικονομία. Θεωρούμε ότι οι επιλογές που έχουν κάνει είναι εγκληματικές γιατί εποάζουν το αυγό του ναζισμού και την άνοδο του φασισμού, αλλά μπροστά στην ανάγκη να υπάρξει ένα στεγανό να αντιμετωπιστεί η επέλαση του φασισμού και ο φασιστικός κίνδυνος, δεν διστάζουμε να βρεθούμε ε, μέσα στα θεσμικά πλαίσια ε, αρρωγή σε προσπάθειες να εφαρμοστούν οι νόμοι, να προασπιστεί η δημοκρατία, να θωρακιστούν οι θεσμοί και να αντιμετωπιστεί ο φασιστικός κίνδυνος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.